Θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτα-πρώτα, γνωμοδότηση Μπαρτ Stars. Θα ψηφίσουμε με ανάταση της χειρός. Ξεκινούμε. Πρώτη τροπολογία για τη λογική 3α. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Μπορεί να τι ψηφίσουμε όλε μαζί, λέει ο κ. Μπέρμαν. Μέχρι πού, από το 1 μέχρι το 4, τι 4 πρώτε. Και τη 10. Επομένως θα κάνουμε μια τροπολογία από το 1 μέχρι το 10. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Εγκρίνεται. Οι πέντε καταπίπτει. Τροπολογία 11 υπέρ. Qui est contre, qui s'abstient, adapté. Εγκρίνεται. 12. Qui est pour? 12 υπέρ, κατά. Qui s'abstient, adapté. Εγκρίνεται. 8. Qui est pour? Οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρώτη συμβαστική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το εννέα έχει αποσυρθεί, οι άλλε καταπίπτουν, επομένω ψηφίζουμε για το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά. Εγκρίνεται. On vote euh, sur le rapport euh, Έκθεση Jolie όσον αφορά το έργο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης ίσης εκπροσώπησης. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πέντε. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έξι. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επτά. υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Όχι. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 7. Ξαναψηφίζουμε. Ανάταση χείρος 7. Υπέρ. 10 είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Εννέα είναι κατά. Και αποχές. Επομένως εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δώδεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε όλες μαζί τις υπόλοιπες. όχι καλά 13 και 14 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 και 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και η παριθμόν 1 πόγκα Τώρα, το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ah, ah, c'est bon, 15. ΑΕΠ έκθεση Ντέβα. Τροπολογία 1. Είναι κάτι το πάρα πολύ ασυνήθιστο, αλλά εάν συμφωνείτε να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 1. Εκεί που λέει τονίζει ότι τα μέτρα, τα οικονομικά δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την, ε, ε, την ανάπτυξη. Και συμφωνώ με, μέχρι να φτάσουμε εκεί που λέει δίκαιη. Μπέρμαν, αγαπητέ συνάδελφε, δεν θέλεις να υπάρχει δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Αυτό λες, λέει ο κύριος Μπέρμαν. Συμφωνείτε να γίνει χωριστή ψηφορία. Κανείς δεν έχει ένσταση, επομένως προχωρούμε και φτάνουμε εκεί που λέει δίκαιη κατανομή εισοδημάτων. Το πρώτο κομμάτι. Τι είναι υπέρ. Δεν συμφωνούν με τη χωριστή ψηφορία οι σοσιαλιστές, άρα δεν θα γίνει. Πρώτη τροπολογία, όπως προήλθε από την κυρία Κέλλερ, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Ζαμπόρσκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5, 6, 7 και 8. Α, όχι, μέχρι το 7. 5 με 7 από κοινού. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η εννέα αποσύρεται. Για το σύνολο της ε, ε έκθεσης. Όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Και δεν θα ψηφίσουμε το ψήφισμα για την Αφρική. Ωραία. Για το σημείο τώρα 16. Ce matin, ont décidé. Αποφάσισαν το πρωί συντονιστές να μην κατεβάσει ψήφισμα η Επιτροπή μας πριν τη συνάντηση κορυφής. Και το μόνο κείμενο το οποίο ισχύει είναι αυτή η κοινή δήλωση Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ε, συμφωνήθηκε. Όμως, αντιθέτως, οι πολιτικές ομάδες πρόκειται να υποβάλουν ένα ε, ψήφισμα για τα συμπεράσματα της συνάντησης του Στρασβούργου. Το Δεκέμβριο θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων, στο Στρασβούργο θα παρουσιαστεί αυτό το κείμενο και πάμε τώρα στο σημείο 17 που είναι η Εθελοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κονγκό σχετικά με την επιβολή δασική νομοθεσίας που διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το νομοθετικό μέτρο που ονομάζεται FLECT. Το άρθρο 81 του κανονισμού προβλέπει ότι όσον αφορά την έγκριση μιας συμφωνίας έχουμε συνολική ψήφιση χωρίς τροπολογίες. Επομένως, θα ψηφίσουμε το σύνολο αυτής της συμφωνίας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Έχουμε ομόφωνη έγκριση. Ακριβώς το ίδιο θέμα τίθεται όσον αφορά την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ένωσης και Καμερούν. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι κατά. Εγκρίνεται. Δέκα είναι. έκθεση της αντιχώρα αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, σύνοδο του ΟΗΕ. Την συνάντηση υψηλού επίπεδου για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Τον Σεπτέμβριο, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, αποτελούμενη από έξι μέλη της Επιτροπής μας, συμμετέσχε στην συνάντηση αυτή του ΟΗΕ σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας γιατί όλοι λάβει δηλαδή, την σχετική έκθεση της αποστολής στη Νέα Υόρκη και θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μίτσελ που ήταν ο επικεφαλής της προσωπία μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την έκθεση. Θα δουν οι συνάδελφοι ότι στην έκθεση όλη την προσωπία ασχολήθηκε εντονότατα και δούλεψε εντατικά για τα πιο πολλές πτυχές ε, τι Συνόδου. Δεν θα σας καθυστερήσω γιατί το συζητήσαμε και στους συντονιστές άλλωστε, αλλά η αντιπροσωπεία αναγκάστηκε να σφίξει τα δόντια για να έχουμε πρόσβαση στην Ολομέλεια, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα για την Επιτροπή εκεί. Ελπίζουμε να επιληθεί. Δεν καταλαβαίνει γιατί ο Επίτροπο Πίμπαλξ αρχικά μάλλον η αίτηση του, το αίτημα του κυρίου Πίβαλξ, του Επιτροπού Πίλβαξ δεν έγινε δεκτό. Ένας από τους ε, συναδέλφους δεν κατάφερε να μπει στην πλατφόρμα, αναγκάστηκε να μείνει απ' έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε κάποια βελτίωση. Θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοι ότι ήταν σημαντικό να βρεθούμε εκεί. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που πήγαμε. Και, να, και το γεγονός ότι πήραμε μία εντύπωση για τις έντονες συζητήσεις, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τους βουλευτές που προσπαθούν να προωθήσουν τους σκοπούς τους. Η Επιτροπή διαβίβασε ένα έγγραφο, δεν ξέρω αν το έχουν όλοι οι βουλευτές, και ανέφερε κάποια από τα επιτεύγματα που έχουν επιτευχθεί. Είναι σημαντικό αυτό, ξέρετε, γιατί ο κόσμος χάνει την ελπίδα του, απελπίζεται. Αν διαπιστώνει ότι δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Όχι λοιπόν, πετυχαίνουμε, έχουμε επιτεύγματα να επιδείξουμε. Φυσικά μπορούμε να καταφέρουμε και πιο πολλά. Και αυτό που πρέπει να καταφέρουμε σε ό,τι αφορά τους στόχους χιλιετίες είναι να κάνουμε ένα sprint, αν θέλετε, μέχρι το 2015. Πρέπει να ανανεώσουμε τις δεσμεύσεις μας και να κάνουμε αυτό το sprint. Να πω ότι ήταν μεγάλη μου τιμή που προέδρευσα της ε, αντιπροσωπείας αυτής και όλοι οι συνάδελφοι έδρασαν με, εξαιρετική, με εξαιρετική συναδελφικότητα και επίσης νομίζω ότι ο κύριος Ντέβα ανάφερε κάποια στοιχεία πριν φύγουμε από τις Βρυξέλλες. Ήταν καλή έκθεση, άξιζε τον κόπο και εμένα να σας πω ότι μου ενίσχυσε την άποψή μου ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας αν επιμείνουμε. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να τα θεραπεύουμε πιο έντονα και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. I'm very pleased to welcome to our meeting our colleagues from the Parliament. Να καλωσορίσω στη συνάντησή μας τους συναδέλφους από, την, ε, από το Κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής. Βρίσκονται εδώ για την 16η διακοινοβουλευτική συνάντηση μεταξύ του Κοινοβουλίου της Νητίου Αφρικής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προεδρεύσει ο συνάδελφος Μάικλ Κάσμαν. Να ευχηθώ λοιπόν μια ευχάριστη παραμονή στους συναδέλφους μας από την Νότια Αφρική και ελπίζω να θεωρήσετε τις συνεδριάσεις μας ενημερωτικές αλλά και ευχάριστες. I now give the floor to Mr. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που καλωσορίζουμε εδώ τους συναδέλφους από την Νοτιοφρική. Με επικεφαλή στην κυρία Φάμπς, με την οποία έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Χαίρομαι που θα μιλήσω για την σύνοδο για τους στόχους της χιλιετίας. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Μίτσελ αναφορικά με την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα της αντιπροσωπείας μας. Συνεργαστήκαμε από όλο το πολιτικό φάσμα, η συνεργασία ήταν καλή. Και ο κύριος Μίτσελ είπε ότι έπρεπε να σφίξουμε τα δόντια για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση και καλύτερο κύρος αν θέλετε. Δεν σφίξαμε τα δόντια. Ο κύριος Μίτσελ απλά ε, ε, ήταν πολύ άκαμπτος και σταθερός και όλοι τον υποστηρίξαμε, διαπιστώνω με χαρά, στην Επιτροπή στη Νέα Υόρκη. Και γι' αυτό λοιπόν καταφέραμε να συμμετάσχουμε στην ε, Ολομέλεια. Οι παράπλευρες εκδηλώσεις ήταν εξαιρετικές και νομίζω ότι άξια εκπροσωπήσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο ενδεχομένως να ενδιαφέρει και τους συναδέλφους από την Νότια Αφρική. Το στάτους το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις, στον ΟΗΕ. Καθόμαστε πίσω-πίσω ως παρατηρητές. Καθόμαστε μεταξύ των διεθνών οργανώσεων για την μετανάστευση και για την κοινοπολιτεία. Και έγινε ένα θέμα, έγινε μια διαδικαστική πρόταση για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, αλλά δυστυχώ πολλοί συνάδελφοι από τις χώρες ΑΚΕ ψήφισαν κατά τις θέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό αίτημα. Άρα δεν συζητήθηκε το στάτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο θα πρέπει να συζητηθεί αυτό, θα πρέπει να είναι πιο έντονη και πιο καλή η εκπροσώπησή μας στο Συμβούλιο. Και αυτό γιατί είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας, ενίσχυσης. Αν δεν λαμβάνουμε εμείς τον εαυτό μας σοβαρά, ποιος θα τον πάρει στα σοβαρά. Το έγγραφο το οποίο προέκυψε είναι καλό, συμφωνώ με τον κύριο Μίτσελ. Και η ανακοίνωση του ε, επιπλέον ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έγινε ε, αποδεκτή με ενθουσιασμό. Αλλά δεν δέχομαι το γεγονός ότι κάποιες ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι ε, παραπονιούνται ότι τα χρήματα αυτά ήδη ήταν στο Ταμείο Ευρωπαϊκής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ευχαριστήσουμε τους δωρητές και να τους δώσουμε περαιτέρω κίνητρα. Το έγγραφο τώρα το οποίο προέκυψε ε, επαναλαμβάνει τα θέματα και τις αρχές καλής διακυβέρνησης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για τις κόκκινες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις. Χαίρομαι λοιπόν που τα πετύχαμε αυτά και χάρηκα που είδα και τη δέσμευση του κυρίου του Πρόεδρου Σαρκοζή. Ελπίζω να τηρήσει τις δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά και τον φόρο των ε, συναλλαγών, χρηματοοικονομικών συναλλαγών και επίσης ε, τις δεσμεύσεις της ε, Άντζελα Μέρκελ. Γιατί όπως ξέρετε και το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και με την κυβέρνηση συνασπισμού, ανέλαβε τις ίδιες υποχρεώσεις. Θα πρέπει λοιπόν σε ό,τι αφορά τον φόρο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών να το θέσουμε στις προτεραιότητές μας το θέμα αυτό. Τέλος, το γεγονός ότι ήμασταν εκεί έδειξε και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και στην κυβέρνηση και στις κυβερνήσεις ότι παίρνουμε πολύ στα σοβαρά το ρόλο μας στον ΟΗΕ. Ήταν εξαιρετική δυνατότητα και ευκαιρία για τον σχηματισμό δικτύων. Δεν έγιναν εκδηλώσεις με ποτό, αλλά πολλές φορές ε, κάναμε τέτοιες επαφές στους διαδρόμους και ήταν εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε τέτοιες διασυνδέσεις. Και έτσι λοιπόν θέσαμε θέματα τα οποία μπορεί να μην είχαμε θέσει αλλιώς. Τα έκανα αυτό και με τον ε, πρόεδρο Καγκάμι από τη Ρουάντα και με τον πρόεδρο Αμπτουλά από την Τουρκία. Του μίλησα τουρκικά και μου απάντησε και αυτός. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι το γεγονός ότι πήγαμε εκεί, ότι καθίσαμε στην ουρά για να πάρουμε τα διαπιστευτήριά μας. Αυτό φυσικά για μένα δεν είναι ιδιαίτερα περίεργο, αλλά για άλλου ίσω να ήταν περίεργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κάναμε. Ο κύριο Μίτσολ μα εκπροσώπησε. Θέλουμε στο μέλλον να έχουμε μπάτς ταυτότητες που να λένε ε, ότι είμαστε βουλευτές, όχι ότι είμαστε σύμβουλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ε, καλωσόρισε θερμότατα και ο Επίτροπος ε, Πίμπαλξ και ο Πρόεδρος Βαρόσο. Έχουμε λοιπόν μια πλατφόρμα επί της οποίας μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για το έργο τους, για την υποστήριξη που μου επέδειξαν ως εισηγητή του Κοινοβουλίου για τους στόχους της χιλιετίας. Και κλείνοντας να πω το εξής. Ένα από τα πιο μία από τις πιο εντυπωσιακέ συναντήσεις που είχαμε, η οποία ξεκίνησε κάπως απεσιόδεξα, γιατί μας ε, ανέφεραν Ήταν τον Τόμα Στέλτσερ από το UNDP, ε, από την ε, Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίο ε, μα είπε, λέγεται, την αλήθεια, όχι αυτά που θέλαμε να ακούσουμε, και μα είπε ότι για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε σε ό,τι αφορά τα ODA θα χρειαστεί στροφή 360 μοιρών. Δηλαδή, αν δεν αντιμετωπίσουμε την επιστηστική ασφάλεια, μα είπε, και την ε, αλλαγή του κλίματος, δεν θα πετύχουμε ποτέ τους στόχους μας. διασυνδέσει όλα τα θέματα τα οποία πραγματευόμαστε, αλλά τα οποία κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, αγνοούμε και αφήνουμε κατά μέρος. Αναφέρθηκε λοιπόν, Πρόεδρε, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τον ακούσει. Να ακούσει ποιε ιδέε έχει να προτείνει αναφορικά με μια πιο συνολική προσέγγιση του θέματο. Θα ήταν λοιπόν σωστό και καλό να τον προσκαλέσουμε στο Κοινοβούλιο. Θα ήταν ωφέλιμο και για τον ίδιο για να συνειδητοποιήσει την δέσμευση υπάρχει στην Επιτροπή μας για την επιτεύξη των στόχων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Νιτον Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κι εγώ είμαι στη μικρή αυτή αντιπροσωπεία και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι δύο συνάδελφοι. Μια πολύ αποτελεσματική, αρμονικά συνεργαζόμενη μικρή αντιπροσωπεία. Το μήνυμα που εγώ συγκράτησα είναι πόσο σημαντική είναι η Ένωση για τα Ηνωμένα Έθνη. Όπως ο Μάκλον, είμαστε του πιο μεγάλους δωρητές και τα κράτη-μέλη πληρώνουν για να, λειτουργεί, να λειτουργούν τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη χρειάζονται την Ένωση και διερωτώ με ο λόγο για τον οποίο ο Γενικό Γραμματέα ήρθε εδώ και μα επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Δεν το είπε. Μήπω έχει σχέση με αυτό. Για την ε, αίτηση, την υποψηφιότητά μα. Ρώτησα υπαγγείλου και έμαθα ότι πήγε από την Νέα Υόρκη στο Ραμπάτ και επειδή είχε απεργίε βέβαια στη Γαλλία και μετά ήρθε στο Στρασβούργο και μετά γύρισε πίσω στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή έκανε μια ειδική προσπάθεια να έρθει να μα δει. Πιθανώς για να ενισχυθεί η θέση μας στα Ηνωμένα Έθνη. Η διαδικαστική ψηφοφορία πριν φτάσουμε εκεί είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν ότι η Ένωση είναι σημαντική, αλλά δεν είμαστε έθνος, αν δεν είμαστε κομμάτι των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε παρατηρητής, είμαστε κάτι μοναδικό, κάτι το ενδιάμεσο. Ο Επίτροπος ζήτησε να ενισχυθεί το καθεστώς μας. Με 76-71 απορρίφθηκε η πρόταση. Και όπως είπε ο Μάικλ και ο Γκέιλ, μόνο έξι χώρες εκεί μας υποστηριξαν, οι άλλες ψήφισαν κατά. Η Αιτή, το Πακιστάν ήταν κατά. Πάρε τα λεφτά που τους δίνουμε. Αλλά ήταν ε, διαδικαστική αυτή η κίνηση. Η τελική ψήφος για το τελικό καθεστώς θα γίνει το Νοέμβριο. Η κάθε άστον που τη συναντήσαμε μας είπε ότι θα φροντίσει την επόμενη ψηφοφορία να την κερδίσουμε τον Νοέμβριο. Αναγνωρίζετε λοιπόν οι, οι αξίες μας. Κι άλλο ένα ανέκδοτο. Ο αναφέρθηκε στο networking με την Προεδρία και είπε ότι συνάντησε κάποιον που νόμιζε ότι ήταν ο Πολ Σμιτ, Ούγκρο Ευρωβουλευτή. Όχι, λέει, είμαι πρόεδρο τη Ουγγαρία, μα είπε. Είμαι πρόεδρο τη Ουγγαρία, δεν είμαι πια ευρωβουλευτή. Τι κάνει εδώ, Είμαι πρόεδρο τη χώρα μου, μα είπε. Α, ωραίο ανέκδοτο. Ευχάριστο. Κάτι άλλο. Το τελικό κείμενο της διάσκεψης ήταν σχετικά ικανοποιητικό, αλλά σχετικά με το θέμα της ευθύνης για τις χώρες που παίρνουν τη βοήθεια, είναι ασθενές αυτό το σκέλος της ευθύνης. Η Ευρώπη θέλει να αναφέρουν οι χώρες αυτές πού πάνε τα λεφτά. Και η εντύπωσή μας είναι ότι θα πρέπει να πιέσουμε για το θέμα αυτό ευθύνης και περισσότερες εξηγήσει πού πάνε τα χρήματα που δορίζουμε. Και το τελικό μου σχόλιο, ένα στέλεχο των Ηνωμένων Εθνών, ο Τόμο, νομίζω, είπε ότι τα Έθνη δεν μπορούν να εφαρμόσουν τι υποσχέσει που δίνουν οι κυβερνήσει. ή υπόσχονται στου δωρητέ ότι θα κάνουν αυτό και εκείνο, γύριζουν πίσω και δεν το κάνουν λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τα Ηνωμένα Έθνη ε, δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν την εφαρμογή αυτών των υποσχέσεων, αλλά μα είπε κάτι άλλαξε. Στα Ηνωμένα Έθνη μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την ισχύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών, emails, κινήσεις λόμπι να πιεστεί η κυβέρνηση να τηρήσει την υπόσχεσή τη. Μεγάλη αλλαγή αυτή. Οι κυβερνήσεις να τηρούν τις υποσχέσεις τους. Και εγώ έφυγα πολύ αισιόδοξο από την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διάσκεψη. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον γειτοντά και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθούμε το καθεστώ. Μια χειραψία με τον Μάικελ και δεδομένη η προαγωγή. Σοβαρά τώρα. Εκεί που σταμάτησε ο Νιούτον Ντάν, τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την τήρηση των υποσχέσεων. Και αυτό αυτός είναι ο κόμπος Υπάρχουν κυρώσεις όμως, οι κυρώσεις της κοινή γνώμης, αν οι υποσχέσεις που ανάλαβε η Ένωση τηρούνται, τότε έχουμε κύρωση στη διάσκεψη. Αν όχι, δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση διαφάνειας έναντι των κρατών μελών, των βουλευτών και της κοινή γνώμης του κόσμου. Και το ερώτημα που θέτω είναι σε τι βαθμό η απόκληση σε σχέση με τις, υποσχέσεις ευθύνεται για την μη υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας και επιπλέον σε τι βαθμό οι υποσχέσεις το να αυξηθούν οι δαπάνες του προπολογισμού της Ένωσης που αποτελεί κομμάτι της ομοφωνίας στην Ένωση για την ανάπτυξη ήταν υπεύθυνη για την μη υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Θα μπορούσε κανείς να πει ό,τι να είναι, ότι δεν μπορεί η Ένωση, δεν με νοιάζει. Αν εμεί θέλουμε οι άλλοι να κινηθούμε στα πλαίσια των εθνών θα πρέπει να είμαστε άψογοι. Και αν είμαστε άψογοι, τότε μπορούμε να παίξουμε το ρόντο αρχηγού σε τέτοιου είδους διασκέψεις. Η επιτυχία μας έχει ένα τίμημα και πρέπει να είμαστε ε, έτοιμοι να πληρώσουμε αυτό το τίμημα. Ο κύριος Ντέβα. Σας ευχαριστώ. Αναφέρθηκε το ότι σαμποτάρισα την διάσκεψη γιατί δεν παρέστην επίτηδες δεν πήγα και νομίζω ότι βοήθησα με την απουσία μου του συναδέλφου που πήγαν εκεί και έτσι αναγνωριστήκε περισσότερο η πρόσφορά του με μεγάλη μου χαρά και εγώ διαπίστωσα ότι πήγε πάρα πολύ καλά η διάσκεψη ήταν ένα επίτευγμα θα θυμάστε ότι ήμουν υποψήφιο για να διαδεθώ τον Κόφη Ανάν ω Γενικό Γραμματέα. και δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα γιατί ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα και ήθελα να γίνω και ο γραμματέας για να το αλλάξω. Συνάντησα τον Μπανκιμούν και συζητήσαμε και τον είχα υποστηρίξει. Όταν κατάλαβα ότι εγώ δεν έχω πιθανότητες να εκλεγώ. Τέλος πάντων θέλω να σας πω ότι δεν πειράζει το τι γράφει η ετικέτα που φοράει κανείς είτε λέει βουλευτής, είτε λέει κάτι άλλο αν κανείς έχει έγχρωμη ετικέτα, πάει στην Ολομέλεια. Ε, αν έχει πράσινη μπορεί να μιλήσει, να λάβει το λόγο στην Ολομέλεια. Αλλά ε, μόνο συγκεκριμένα χρώματα ετικέτας ε, επιτρέπονται στην Ολομέλεια. Αυτό ήθελα να σας πω. Τα είπαμε στην Επιτροπή και μου απάντησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν του τα είπα. Τα εσείς με τους συντονιστές. Και είπε ότι όλα πήγανε πάρα πολύ καλά και λοιπά και λοιπά. Τον συνάντησα στο αεροπλάνο και μου έκανε τον καλό. Αλλά τέλος πάντων έτσι θα έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Έτσι θα έπρεπε να κάνω. Τα έχω κάνει αυτά πολλές φορές και ήταν η συμπεριφορά απέναντί μου πάρα πολύ άσχημη. Όμως θα πρέπει ο ΙΕ να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη πέραν εξωτερική πολιτικής. Αλλά όσον αφορά τα θέματα ανάπτυξης, εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής και δεν είναι δυνατόν να μας μεταχειρίζονται σαν να είμαστε σκουπίδια. Γι' αυτό και μίλησα στο Γενικό Γραμματεία και σε άλλους από την γραμματεία του Γενικού. Επομένως, δεν θα πρέπει να μείνουμε ε, στο θέμα αυτό σαν ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Δεν είναι ένα απλό τέτοιο θέμα. Ε, δεν είναι μια σκιά με την Επιτροπή. Θα πρέπει να δώσουμε θεσμικό, χαρακτηριστικές διαστάσεις στο θέμα αυτό γιατί ο κύριο Μίτσο και ο κ. Κάσμα τα πήγαν πάρα πολύ καλά, γίνανε θεσμικά βήματα πρόοδου. Θα πρέπει αυτό επομένω να αξιοποιηθεί. Δεν ξέρω ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία, αλλά κάποιο θα πρέπει τώρα να πει ότι στο μέλλον έτσι θα προχωρούμε. Ακόμα και ένας μόνο βουλευτής να πηγαίνει στον ΟΗΕ να παίρνει την ετικέτα, το μπάτζ αυτό, το κόκκινο, για να μπορεί να μπει στην συνέλευση. Κύριε Γκερέρο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από αυτά που μας είπαν οι συνάδελφοι ότι για την προσωπία μας που απεστάλλει εκεί τα πήγε πάρα πολύ καλά όσον αφορά του στόχου της χιλιετία. στις επίσημες ε, εκδηλώσεις, στις συναντήσεις, στις ε, εκδηλώσεις της παράλληλες που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αυτής της διάσκεψης. Και το αποτέλεσμα, ακριβώς όπως αναφέρει το τελικό έγγραφο, αλλά και όσον αφορά τα όσα συμφωνήθηκαν ε, από θεσμικούς παράγοντες ή από εκπροσώπους της κοινωνίας ή επαγγελματικών κύκλων μπορεί να μην είναι πλήρως ικανοποιητικό αλλά τουλάχιστον δίνει κάποια αισιοδοξία ότι δηλαδή σε μια συγκυρία τέτοια κρίσης που αφορά και την αναπτυξιακή βοήθεια μια λοιπόν που έχουμε αυτή την χρηματοοικονομική κρίση και αυτό απειλεί την ανάπτυξη των φτωχών χωρών, οι περισσότεροι εμπλεκόμενους τήρησαν τα υπεσχημένα. Και αυτό ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, μάλιστα ανελήφθησαν επομένω και νέες ε, υποχρεώσεις όπως αυτό το εκατομμύριο των ευρώ που υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπε ο κύριος Γκέρενς, θα πρέπει να τηρούμε 100% τόσο έχουμε υποσχεθεί μια που ακριβώς είμαστε ο βασικός δωρητής και να είμαστε ένα παράδειγμα προς ε, μίμηση για τις ανηλυμένες υποχρεώσεις μας που τηρούμε και ο Μάικλ Κάσμαν που προβληματίζεται όσον αφορά την κυβέρνηση της... Ε, και μάλιστα έκανε για το λάθος, Η κυβέρνηση σύγκρουση και όχι συνασπισμού. Ε, γλώσσα λανθάνουσα. Οπότε θα, το, το παραπέμπω σε εκείνη την ε, δήλωση του, του Ισπανού Πρωθυπουργού όσον αφορά τη φορολόγηση των ε, χρηματιστηριακών συναλλαγών. Και έχουμε επομένω κρίση δημοσιονομική, κρίση απασχόληση στην Ισπανία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι συνεχίζεται η πολιτική της αναπτυξιακής βοήθειας. Σε τέτοιες συνθήκες. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Κάσμανος, στον αυρό θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε για ένα πιο συνολικό όραμα, πιο συνολική οπτική και για κάποια άλλα μέσα πολιτικής ευρύτερα όσον αφορά τα προβλήματα της ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015. Μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον προβληματισμό η Επιτροπή μας. Θα είναι πολύ θετικό. Τέλος. Η επόμενη συνάντηση των G20 θα γίνει στη Σεούλ. Και στην ημέρα διάταξη υπάρχει ένα σημείο προς συζήτηση που αφορά την ανάπτυξη. Και είναι πρώτη φορά που οι G20 θα συζητήσουν την ανάπτυξη. Αυτό έγινε τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα θα ήταν μια καλή ιδέα. Η Επιτροπή μας, ίσως μέσω κάποιας δήλωση ε, της Προέδρου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να τοποθετηθούμε υπέρ του να συζητηθούν ουσιαστικά στη Σεούλ τα θέματα της ανάπτυξης και όχι απλώς να είναι ένα σημείο στη μέση διάταξη. Να είναι εκεί ως σημείο ε, σημαντικό για τις ε, ευκαιρίες, τα δεδομένα που μπορούν να ε, έχουν σημασία για την ανάπτυξη την παγκόσμια την επόμενες δεκαετίες. Πρόεδρος. Κάσμαν και Ντέβα. Έχετε ο καθένα από ένα λεπτό για να δευτερολογήσετε. Λιγότερο από ένα λεπτό να απαντήσω στα σχόλια του κύριου Γκέρεν. Έχει δίκιο. Με τι υποχρεώσει αυτέ, αν δεν υπάρχουν κυρώσει και εξοχιστικός έλεγχο. δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Βέβαια, η Ισπανική κυβέρνηση όντω σωστά έχει αναλάβει μια δέσμευση. Η Επιτροπή μα. θα πρέπει να κάνει μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία ετήσια όπως θα παρακολουθούμε το κατά πόσον οι δεσμεύσεις των κρατών μελών υλοποιήθηκαν. Αυτό ήταν καλός τρόπος για μας να παίξουμε ηγετικό ρόλο, γιατί ακόμα και με το τελικό έγγραφο δεν υπάρχει εξοχιστικός έλεγχος και παρακολούθηση. Και με τη θέση της Ένωσης πάλι κάτι λείπει. Αυτό είχα να προτείνω. Και ο κύριος Ντέβα. Ο κύριος Γκέρνς ε, με υποχρεώνει να σα θυμίσω τα καλά νέα από την Αγγλία. Όταν περικόπη ο προπολογισμό την περασμένη εβδομάδα κατά 25%, ο προπολογισμό για την ανάπτυξη αυξήθηκε κατά 37%. Θα έχουμε το στόχο του 0,7% του ΑΕΠ και η δέσμευση αυξήθηκε κατά 4,8 στερλίνες δις στερλίνες το χρόνο. Δηλαδή κόβουμε τις υπηρεσίες τους Βρετανούς, σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Ίσως όχι ακόμα, πάντως Ωραία, προστατεύονται τα νοσοκομεία. Τα σχολεία, ας πούμε, θα κλείσουν ορισμένα σχολεία. Αυξάνουμε τον προπολογισμό ε, ανάπτυξη κατά 37%. Και τώρα το λόγο στην επικεφαλή Επικεφαλή της αντιπροσωπείας από την Νότια Αφρική, την κυρία Φίμψ. Έχετε μερικά λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μας να ακούσουμε έστω και λίγο από αυτό που κάνετε θα μια μεγάλη ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις εργασίες της δικής σα Επιτροπής και άλλων Επιτροπών και που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο. Στη Νότια Αφρική μας ενθαρρύνεται να βλέπουμε του αυτούς μας σε ένα κομμάτι μιας ευρύτερης περιοχής της Αφρικής. Γνωρίζουμε τη βοήθεια που την έχουμε μοιραστεί με χώρες της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης και της Νότιας Αφρικής. Αλλά θέλουμε να το εκφράσουμε και σε εσάς ως Επιτροπή την ανάγκη για αυξημένη βοήθεια σε τομείς κλειδιά, όχι μόνο για διακυβέρνησης για ειρήνη και ασφάλεια και οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την την τεχνολογία, τεχνολογική ενίσχυση. Ταυτόχρονα εκτιμούμε το ότι ήδη συμβάλλεται και προς την Νότια Αφρική για ένα πρόγραμμα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και ήδη στέλνετε βοήθεια, όπως μέχρι και πρόσφατα ανεφέρθηκε προς τον πρόεδρο Ζούμα ότι αυτή η βοήθεια, βοήθεια για τα δημοτικά σχολεία και ότι είναι ευπρόσδεκτη η βοήθεια αυτή της Ένωσης. Και η εταιρική μας σχέση έχει ιδιαίτερη αξία για μας, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς, κυρία μου. Η Κομισιόν τώρα. Ο κύριος Χαρ Πολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε και εμείς με αυτά που είπαν οι ευρωβουλευτές ότι η διάσκεψη υπήρξε επιτυχία και όσον αφορά τα έγγραφα και όσον αφορά τη συμμετοχή με 110 επικεφαλής κυβερνήσεων και κρατών και πολλοί από αυτούς δεσμεύτηκαν δημόσια. Μια θετική ορμή λοιπόν εξασφαλίστηκε. Τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε όλα αυτά να εφαρμοστούν. Η Ένωση έπαιξε το ρόλο της και με την καλή προετοιμασία που είχε κάνει ε, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Κομισιόν, το ιερνό πακέτο, τα απορίσματα του Συμβουλίου, η δουλειά του Κοινοβουλίου, η δουλειά του κ. Κάσμαν με την ε, φροντίδα των ε, νηπίων και των ε, ε, μητέρων. Η σημασία της Ένωσης να τηρήσει τη δέσμευση του 0,7% που ανέφερε ο κύριος και αυτό μέτρησε για τις διαπραγματεύσεις η δημόσια δέσμευση του κυρίου Μπαρόσο με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ταμείου επιπλέον ένα δις και αυτό σαφέ Η συζήτηση στη Νέα Υόρκη τι γίνεται πέραν της βοηθείας. Πράσινη ανάπτυξη, κινητοποίηση εσωτερικών πόρων, παράνομες ε, ροές κεφαλαίων, ο φόρος για τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές πράξεις, όλα αυτά ανοίγουν νέες προοπτικές για νέα εργαλεία και όπως είπε ο κύριος Μίτσελ, χρειάζεται ένα κατοστάρι αυτή τη στιγμή να τρέξουμε και είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Το τελικό κείμενο, 32 σελίδες, 192 χώρες, μοιραίο ήταν αυτό να είναι τόσο μεγάλο, καλό έγγραφο. Το να μην έχουμε έγγραφο θα ήταν κάτι πολύ σοβαρό δεδομένων των δυσκολιών λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κλπ. κρίσης είναι θετικό. Και για τα Ηνωμένα Έθνη ήταν σημαντικό για, την πολυμερή δράση των Ηνωμένων Εθνών. Ας υποστηρίξουμε αυτό που είπαν οι ευρωβουλευτές, το τι είναι επιτεύξιμο και είναι τιμή μου να σας μιλάω σήμερα εδώ και έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα τη σταδιοδρομία σας κύριε Πρόεδρε και το παράδειγμα που δίνετε. Χαίρομαι λοιπόν για το ότι όλοι συμφωνούμε. Πρόεδρος. Ο κύριος Μίτσελ θέλει το λόγο. Ναι, ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πρέπει να φροντίσουμε η ορμή αυτή να μην σταματήσει για να τρέξουμε το τελευταίο αυτό κατοστάρι σε σχέση με το στόχο μας. Και όπως είπε ο κύριος Κάσμαν, έχουμε μια ετήσια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Το σημειώνουμε και αυτό για τη συνάντηση των δωρητών. Περνάμε στο επόμενο. Σημείο 20 μηχανισμός χρηματοδότησης αναπτυξιακή συνεργασία τραγωποίηση του κανονισμού. Το θέμα των νομιμοθετικών αλλαγών που προτείνει η Κομισιόν στο, στο μηχανισμό χρηματοδότησης αναπτυξιακής συνεργασίας, στον κανονισμό ICD. Ο κύριος Μίτσελ είναι για την αναθεώρηση, την ενδιάμεση αναθεώρηση και ο κύριος Γκέρες είναι εισηγητής για την προσθήκη ενός νέου τμήματος συνοδευτικών μέτρων υπέρ των χωρών ΑΚΕ που παράγουν μπανάνα. Θα μελετήσουμε από εκείνου τα σημεία 20 Θα ακούσουμε τους δύο εισηγητές. Τι κατεύθυνση παίρνουν οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν και το Συμβούλιο με βάση την εντολή και τα όρια που όρισε η Επιτροπή μας εγκρίνοντας ομόφωνα αυτές τις δύο εκθέσεις. Πρώτος ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε είμαι συγγητής για την ε, πρόταση τροποποίησης του κανονισμού αυτού για την αναπτυξιακή συνεργασία και σκοπός μας είναι να εισάγουμε ευελιξία για την καταβολή φόρων σε ό,τι αφορά τις χώρες όπου ε, γίνονται δράσεις αναπτυξιακές. Αυτό γίνεται γιατί οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις συχνά δεν έχουν σε θέση να διαπραγματεύονται ε, απαλλαγές, φοροαπαλλαγές. Θέλαμε λοιπόν να εισαχθούν τα μέτρα επιτροπολογίας και τροπολογίες αυτές ε, εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα και έγιναν και κάποιες προτάσεις τον Ιούλιο από την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. η ΑΦΕΤ, η ΙΝΤΑ και η ΔΕΒΕΤ και να υπάρξει και μια ομάδα διαχειριστική με τους προέδρους όλων των επιτροπών. Συμφώνησαν λοιπόν οι επιτροπές ότι θα πρέπει να ψηφιστεί η έκθεση τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια, άσχετα από το αν θα υπήρχε συμφωνία στους στα άλλα όργανα, που δεν υπήρξε τελικά. Και κατά την ψηφοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε κάποιες μικρές τροποποιήσεις της ομάδας εργασίας για να υπάρχει διαβούλευση του Κοινοβουλίου για τα αιτήσια πρόγραμμα, προγράμματα. Παρά το γεγονό ότι ήμασταν πολύ σαφεί για την ψηφοφορία που θα γινόταν τον Οκτώβριο, μία εβδομάδα πριν ε, μας υποβλήθηκε από την, το γραφείο του κυρίου Μπαρόσο το αίτημα να αναβληθεί η ψηφοφορία. Και την ημέρα πριν από την ψηφοφορία έγινε μια συνάντηση μεταξύ των τριών οργάνων και συμμετείχε και ο Επιτροπός Πίβαλξ και η ε, κυρία Άστον καθώς και η Βαλγική Προεδρία η είπατε εκπρόσωπος Άστον δήλωσε στη συνάντηση αυτή ότι δεν υπήρξε πρόταση της Επιτροπής και επέμενε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Είπε ότι θα έπρεπε να γίνουν συναντήσεις μεταξύ του προσωπικού. Έγινε μια συζήτηση την ίδια ημέρα και η θέση της Επιτροπής ήταν ακριβώς η ίδια με αυτήν που μας ε, αναφέρθηκε επανειλημμένα τους προηγούμενους μήνες. Στα ίδια δηλαδή, τα ίδια τόνισαν και σε ό,τι αφορά τις delegated acts και σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλεγχο χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε υποχώρηση σε ό,τι αφορά την επόμενη περίοδο. Και τέλος ζητήθηκε να γίνει εκ νέου διαβούλευση με τα μέλη του Κοινοβουλίου για την πρόταση αυτή. Και θα ήθελα να τονίσω το εξή, επειδή ήμουν παρόν, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Απορρίπτω μια λύση η οποία δεν ε, περιλαμβάνει πράξεις κατανάθεσης. Είμαστε συνομοθέτης. Δεν είμαστε μια απλή ένωση. Κατά δεύτερον, δεν ε, δέχομαι μία ενδιάμεση λύση γιατί θα αποτελέσει προηγούμενο για το μέλλον. Τώρα θα πρέπει να τα λύσουμε τα θέματα και πάντα αυτή ήταν η θέση της θέσης ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της διάσκεψης των Προέδρων και μετά την τελευταία ψηφοφορία και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, Πρόεδρε, όσο εφόσον θα περάσουμε στην δεύτερη ανάγνωση, ελπίζουμε να προχωρήσει η συζήτηση, να μην ε, μείνει η Επιτροπή στα επιχειρήματα του παρελθόντος. Καταλαβαίνουμε ότι έχει αυτή τη θέση της, αλλά να συζητήσουμε μόνο εφόσον υπάρξουν κάποιες νέες προτάσεις, γιατί ο Πρόεδρος Μπαρόσο μας είπε ότι προετοιμάζει μια νέα πρόταση. Να τη δούμε λοιπόν. Αν μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας νέας συμφωνίας γιατί ο μοναδικό τρόπο να προχωρήσουν τα μέσα αυτά είναι αν κάτσουμε και συζητήσουμε στα σοβαρά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Και τώρα ο κύριο Γκιόρεντ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ έχω αναλάβει μια έκθεση κατόπιν τη ψήφισή όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα για την ε, μπανάνα. Στις 6 Οκτωβρίου μου αναθέσατε την διαπραγματευτική εντολή ως προς Κομισιόν και Συμβούλιο για την έκθεση όσον αφορά αυτά τα συνοδευτικά μέτρα για την Πανάνη. Ούτως ώστε να αναλυθεί ένα μέτρο νοτιακή βοήθειας και εδώ έχουμε μια δέσμη μέτρων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις 10 ε, χώρε παραγωγές της ε, ΑΚΕ. Εγκρίθηκε στην Ολομέλεια η έκθεση 574 ε, ψήφους υπέρ. Οι περισσότεροι από εκείνους που δεν υπερψήφισαν ήταν απόντες. Πάρα πολύ λίγοι κάτε ψήφισαν τώρα όσον αφορά τα σχετικά μέτρα. Τελικά συμφωνήθηκαν ακόμα και στα πιο επιμεχά σημεία, όπως η πραγματική κλίδα κατανομής για τις 10 χώρες. Είχαμε επίσης και την ε, Αξιολόγηση, την αναγκαιότητα του να έχουμε σε ψηλή προτεραιότητα το τι θα γίνει με τους ε, χωρικούς τους εργαζόμενους στον κλάδο αυτής της δραστηριότητας. Και τελικά συμφωνήσαμε απόλυτα Κομισιόν και Κοινοβούλιο και αυτό πρέπει σε σχέση με αυτή την υπόθεση να ευχαριστήσω όλου του σκιώδε ηγητέ, ο κύριο Πόγκα, η κυρία Γκρά και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι βοήθησαν με τι παρατηρήσει του, με την ανταλλαγή απόψεων με το θέμα αυτό. Και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά να ζητήσουμε κάποιε λύσει όσον αφορά ε, τον κλάδο αυτών. Και τελικά τα βρήκαμε όπως είπαμε με Συμβούλιο και Επιτροπή. Είπαμε ότι θέλουμε γενικότερα να αναλάβουμε δράση, να εντείνουμε την εξωτερική πολιτική και αυτό είπαμε ότι θα γίνει με τέτοιες κατουσιοδότηση πράξεις και πιο συγκεκριμένα ε, έχουμε το καινούργιο άρθρο 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την νέα στρατηγική ε, οπότε και συνεργαστήκαμε στενά με όλους τους ε, συντάκτες των κειμένων και με την Κομισιόν, τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Σας τα εξήγησε ο κύριος Μίτσελ. Σε πρώτη ανάγνωση επομένω, ε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ήταν η θέση της Επιτροπής μας, αυτή που ε, αποκρισταλώθηκε, τα είπαμε την κυρία Άστον και τον κύριο Πίμπαλτς και έτσι. Πήγαμε στη δεύτερη ανάγνωση όπου θα αναλάβω και εγώ τις ε, σχετικές επαφές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των μέτρων εξωτερικής συνεργασίας δεν θα περιοριστούμε ε, σε μια απλή ε, αρμοδιότητα έγκλησης, αλλά λοιπόν ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε να αλλάξει τη στάση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που θα ξεπεράσει τα όρια των ομοδιοτήτων όπως αυτές ε, προβλέπονται σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε κάποια στρατηγικά έγγραφα για τα συνοδευτικά μέτρα. Αυτό το έγγραφο το εξεπώνησε η Επιτροπή και θα πρέπει να εγκριθεί όπως προβλέπεται για τις κατοξιοδότες πράξεις. Οπότε, όπως βλέπετε, έχουμε τρεις επιλογές. Πρώτα-πρώτα, να πούμε ότι όλα είναι τόσο καλά και δεν λέμε τίποτα. Δεύτερον, να σταματήσουμε την διαδικασία που δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ είμαστε ψηφία και το τρίτον είναι αυτό το οποίο διαπραγματευτήκαμε και αυτό το οποίο μας εξήγησε ο κύριος Μίτσελ με τον οποίο συμφωνώ. Οι δύο πρώτες επιλογές ουσιαστικά οδηγούν στην τρίτη. Όλη η Επιτροπή συμφωνεί και συμφωνώ με τον ε, Γκέι ότι προσωρινές ε, συμφωνίες δεν εξυπηρετούν προσωρινές λύσεις. Χρειάζεται τέτοια κατοξιοδότηση πράξη για όλα τα θέματα που έχουμε να ρυθμίσουμε και για τα συνδευτικά μέτρα και για όλα. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θεωρητικό. Πάρα πολύ θετικό το ότι δουλέψαμε πάρα πολύ, ε, ε, πάρα πολύ, με πάρα πολύ καλή συνεργασία όσον αφορά αυτή την ε, έκθεση και έτσι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε σε μια εύστοχη λύση η οποία κατοχυρώνει τις απόψεις όλων. Merci. Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Γκράση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω εάν θα με προσέξουν όλοι όσο τους προλαλήσαντες, αλλά όντως θα σας πω ότι δουλέψαμε πνεύμα συνεργασίας, αλλά χωρίς να πω στην ουσία θα θέλω να σταθώ σε κάποια στοιχεία Έχω κάποιες ερωτήσεις, έχω κάποια που θέλω να τονίσω. Νομίζω ότι ο ρόλος της Επιτροπής μας είναι πάρα πολύ σημαντικός για αυτό το θέμα, όπως άλλωστε και για άλλα τα οποία αφορούν εμπορικά θέματα. Και γι' αυτό έτσι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις αντισωμένες χώρες και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις τροπολογίες, τι γίνεται με τα διοκτώνα για τα φυτοφάρμακα και ο κύριος Γκέρνς μας έχει προτείνει να γίνει μια έκθεση αξιολόγηση των επιπτώσεων ε, οπότε και εγώ ε, θέλω να δούμε κατά πόσον αυτό είναι εφικτό, με ποια διαδικασία θα καθοριστούν τα κριτήρια αυτής της ε, μελέτης επιπτώσεων γιατί νομίζω ότι αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια μελέτη όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία, τα, το, το, τη χρήση προϊόντων ε, χλωρίου. Όλα αυτά νομίζω ότι μας οδηγούν στο ότι για όλες τις ε, συμφωνίες για την μπανάνα ε, μιλούμε βέβαια για χώρες σακέ, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε τον κλάδο της μπανάνας και ο κύριος Στυρολίου είναι συμφωνία μαζί μου Ε, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις ε, χώρες ΑΚΕ. Γουαδελούπη, επίσης, Μαρτινίκα, γιατί και αυτές οι χώρες είναι παραγωγή μπανάνας. Ευχαριστώ. Ε, je donne la parole à moi-même. Je pense que... Πρόεδρος, θα μιλήσω τώρα εγώ. Ο ρόλος της Επιτροπής μας και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός. Και η Ένωση από την αρχή σιγά σιγά φτιάχνεται προχωρώντας. Έχουμε μια νέα συνθήκη και τη μάχη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και για τη μελλοντική λειτουργία μας. Γιατί οι αντιστάσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Σαν να δίνουν μάχη οπισθοφυλακής. Γιατί το νόημα της ιστορίας μας λέει να ενισχυθεί η δημοκρατία στους θεσμούς μας και να δοθεί στους εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού η δυνατότητα ελέγχου των πράξεων που αφορούν τους συμπολίτες μας. Τι θα γίνει αν δεχτούμε για 7 χρόνια να μην μπορούμε να παρέμβουμε για τα χρηματοπιστωτικά, χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία. Κατ' επανάληψη βλέπουμε τον πειρασμό να ενσωματωθούν στους μηχανισμούς αυτούς και άλλα μέτρα για την ανάπτυξη. Αυτό τον πειρασμό το βλέπουμε και σήμερα. Καθημερινά οι κυβερνήσεις θέλουν το κόστος του ελέγχου της μεταναστευτικής ροής να μπει στις δαπάνες για την ανάπτυξη. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε σε αυτόν τον πειρασμό. Πιστεύω ότι όλοι θα καταλάβουν ότι το συμφέρον είναι το Κοινοβούλιο να μπορεί να ελέγχει αυτές τις πράξεις. Γιατί αυτό είναι το νόημα της ιστορίας. Η θέλει να πει κάτι. Όχι. Το συμβόλιο, ο κύριος Γκύραγε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μίτσερ και τον κύριο Γκέρενς και σας για τη σαφή σας θέση η θέση του Συμβουλίου είναι επίσης σαφής. Γνωρίζετε τη θέση και της Κομισιόν και του Συμβουλίου και των νομικών υπηρεσιών και των δύο υπηρεσιών. Στη συνεδρίαση με τον κύριο Άστον, ο κύριος Πίμπαλς, τον εκπρόσωπο του κύριου Σαστέλ και αποφασίστηκε να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος άτυπα. Η πρώτη επίσημη συνεδρίαση θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου. Θέλουμε κι εμείς να βρεθεί μια ρεαλιστική λύση για τους δύο μηχανισμούς έκθεση Μίτσελ, έκθεση Γκέρνες, δεν έχουμε πρόβλημα στο Συμβούλιο. Ούτε ως προς την ουσία, ως προς το περιεχόμενο των προτινόμενων μέτρων. Είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί η συζήτηση. Στις 20, όπως υπόθηκε από τον εκπρόσωπό μας, στις 20 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο οι συγητέ μας ξανά. κύριο κύριος Μίτσελ πρώτος. Ευχαριστώ. Εγώ και ο συνάδελφος Γκέρενς ακούσατε τη θέση μας. Για να περάσει η συνθήκη της Λισαβόνης χρειάστηκε να περπατήσω πάρα πολύ στους δρόμους του, του Δουβλίνου. Δύο φορές. Με απογοητεύει το γεγονός ότι η Κομισιόν συχνά συντάσσεται με το Συμβούλιο αντί να είναι αμερόληπτη στη στάση της. Και αυτό πρέπει να σταματήσει κάποτε η Κομισιόν. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να συμβάσει τις θέσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ως ουδέτερος μεσολαβητής, όχι μεροληπτικά. Συμφωνήσαμε να επιληθεί αυτό μόνο αν ε, υπάρξει πλήρη σεβασμό των εξουσιών του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε λοιπόν τη συμμετοχή του Συμβουλίου, αλλά είμαστε σαφείς. Το θέμα αυτό δεν θα επιτρέψουμε να παραχθεί. Θα το πρέπει να το χειριστούμε ως όριμοι νομοθέτες. Και ο κύριος Γκέρανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα εμπνευστώ από το ο είπε όποιος έχει εξουσία μπαίνει στον πειρασμό να καταχραστεί την εξουσία. Ποιο στην απόλυτη εξουσία, το ίδιο συμβαίνει. Όταν μοιραστεί την εξουσία με κάποιον άλλον, η πιθανότητα κατάχρηση είναι και αυτή μοιρασμένη. Πρέπει να, να φροντίσουμε να μοιράζεται εξίσου η εξουσία. Παράδειγμα, με τον Κομισιόν, στην ανταλλαγή απόψεων που οδήγησαν στα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα, είχαμε μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Το Κοινοβούλιο δεν σαμποτάρισε Παράδειγμα, το μέτρο όπου καλέσαμε την Κομισιόν να κάνει μία μελέτη επιπτώσεων εκ των προτέρων. Η Κομισιόν παρουσίασε τα επιχείρηματά της, εμείς τα δικά μας, υιοθετήσαμε τα, το επιχείρημα της Κομισιόν και ο συμβασμός ήταν αντί να το πούμε αξιολόγηση εκ των προτέρων για να μην χάσουμε χρόνο για να ισχύσουν τα μέτρα αυτά, συμφωνούμε. Να προτρέξει κατά κάποιο τρόπο η αξιολόγηση, όπως προβλέπετε, πριν τους 18 μήνες, πριν αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα. Αυτός ο συμβασμός, σε αυτόν δώσαμε τη συμφωνία μας και έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη λεπτή περίπτωση θα υπάρξει και εδώ λύση με διαπραγμάτευση για να ενθερθεί η Κομισιόν. Εξάλλου τα στελέχη της Κομισιόν που είναι σήμερα εδώ είναι λογικοί άνθρωποι. Και θα πρέπει η κοινή λογική θα πρέπει να περάσει και προς τους προϊσταμένους τους για να πετύχουμε αυτή τη συμφωνία που όλοι τη θέλουμε. Το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο και εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσία του στελέχους του Συμβουλίου σήμερα με τις σπάνιες ευκαιρίες. Επειδή πολλές άλλες ευκαιρίες συνάντησης και συζήτησης με το Συμβούλιο μας έχουν αφαιρεθεί και λυπάμαι γι' αυτό. <clears throat> Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Περνάμε στο επόμενο σημείο. η συμφωνία για την, ε, το εμπόριο της μπανάνας. δώσουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εμπορίου. Η συγητής μας είναι ο κύριος Γκέρενς. Το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο την έγκριση της συμφωνίας της Μπανάνας μεταξύ της ε, ε, Βενεζουέλας, Κολομβίας, ε, Ουαταμάλα, Κωνσταντίνα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμά, Περού, Βενεζουέλα και μια συμφωνία του εμπόριου της μπανάνας μεταξύ της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών το λόγο και πάει στον κύριο Γκέρνς. Πέντε λεπτά. Δεν μου χρειάζονται πέντε λεπτά. Είναι μια γνωμοδότηση. Αναφέρω τη θέση μας που υπάρχει στην βασική έκθεση για τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι μειώνονται οι προτιμήσεις χωρίς να υπάρχει μια εναλλακτική λύση για τις χώρες που παίρνουν τη βοήθεια. Αυτό, η Επιτροπή Ανάπτυξης μας ενοχλεί. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται, ακολουθεί τις συστάσεις με βάση την ομοφωνία της Ουάσιγκτον θα πρέπει να ξαναδούμε πώς ε, τι γίνεται με αυτή τη μείωση των γενικευμένων προτιμήσεων. Ορισμένες χώρες δεν καταφέρνουν μόνες τους να βγούνε από την αθλειότητα στην οποία βρίσκονται. Γι' αυτό πρέπει να τους ακούσουμε και να αναζητήσουμε τρόπους που θα τους βοηθήσουν να προχωρήσουν προς τα μπρος, χωρίς να εκτίθενται βία σε αλλαγή μιας κατάστασης διότι εμείς στηριζόμαστε σε συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα, για δεσμολογική μείωση 175 ευρώ τον τόνο σε 114 ευρώ τον τόνο στην εισαγωγή στην Ένωση. Μείωση των δασμών αυτό αλλάζει πολύ σημαντικά τη διαφορά που υπήρχε πριν. Πριν, ισχύσει, πριν ισχύσουν τα τρέχοντα μέτρα, προστατευόντουσαν οι χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Σιγά σιγά πάβει να ισχύει αυτό, χωρίς να έχουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν τον βίο αυτό ανταγωνισμό οι χώρες αυτές, παγκόσμια. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια βαθμία λύση έτσι ώστε νέα μέτρα να μην εφαρμοστούν αμέσως. Διότι αυτό που συμβαίνει τώρα και αυτό μέχρι το 2020 προοδευτικά καταργούνται με ορατό τρόπο μέτρα μείωσης των δασμών από 114 σε 75 ευρώ τον τόνο. Και αν εφαρμοστεί η προτίμηση του έθνους του λιγότερο ευνοημένου, του, του πιο πολύ ευνοημένου, θα πρέπει οι χώρες αυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το δεσμολογικό καθεστώς επίπεδο. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Τι θα γίνει μετά το 2013. Δυστυχώς τα μέτρα μας σταματάνε το 2013, γιατί έχουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές που σταματάνε εκεί. Δεν θα έπρεπε όμως το χρονοδιάγραμμα να επιβαρύνει την ουσία. Αυτή είναι η ουσία της έκθεσής μου. Έκθεση γνωμοδότηση Προσπάθησα να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Ελπίζω η Επιτροπή μας να συμφωνήσει με αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Κεράνης. Καλώς όρισαν οι προσκεκλημένοι μας. Ε, σας εύχομαι καλά να περάσετε εδώ στην επισκέψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να σας προσφέρει κατευθείαν αυτή η επίσκεψη. Κύριε Γκέρτζη, έχετε συναντήσει το λόγο. Ναι, ε, ε, εγώ τους έχω καλέσει και είστε ε, πολύ βγαίνει τα λόγια σας και επίσης το πιο, είναι σωστό να βγαίνει προς τα έξω το έργο μας. Αυτό ήθελα να κάνω έστω και έτσι σαν και κροτές, ήθελαν να έρθουν εδώ οι προσκεκλημένοι μου και ε, μόνο έτσι ίσως ε, γίνεται αυτή η προβολή του έργου μας. Κύριε Υπάρχει επικάλυψη μεταξύ αυτών των θεμάτων, οπότε και εγώ θέλω να σα πω πιο συγκεκριμένα αυτά τα οποία με απασχολούν σε σχέση με αυτά που μα είπε ο κύριο Γκέρντ όσον αφορά ακριβώ τη μελέτη επιπτώσεων σε σχέση με αυτή την εμπορική συμφωνία με τις αμφισόμενες χώρες. Επίσης θα πρέπει να εξηγηθεί πώς καθορίζονται τα κριτήρια για την μελέτη της αξιολόγησης των επιπτώσεων. Εμείς πώς μπορούμε να εμπλακούμε και εγώ θα ήθελα να υπάρχει ιδίως όσον αφορά τα παραστοκτονομία μία μελέτη και το τελευταίο μου θέμα είναι ότι πόσο όσον αφορά το εμπόριο της μπανάνας θα καλυφθεί ε, το θέμα ε, Μαρτινίκας, κλπ. Bon. est Πρόεδρος, θέλει η Επιτροπή το λόγο. Μου είπαν ότι είναι τρεις οι αρμόδιοι που παρίστανται. Ο κύριος Βίλεμ Όλτχολ η κυρία Λτρομελής και ο κύριος Λούκος. Thank you, Madam Chair. And, um... Ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για το προηγούμενο θέμα για τα μέτρα για την μπανάνα. Θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στις ερωτήσεις που έκανε η κυρία Γκρέσ. πώς μπορούμε να ενισχύσουμε στις διάφορες χώρες τις στρατηγικές. Μια μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα και τις ε, εργασιακές συνθήκες και το καθεξής. Όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς στη συζήτηση που έγινε μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής και Κοινοβουλίου, προτάθηκαν κάποιες τροποποίησεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτές συγκαταλέγονται και κάποιες τροποποιήσεις για το πώς θα πλαισιωθούν οι στρατηγικές στις διάφορες χώρες. Είναι σαφές στο νομικό πλαίσιο ότι όλες οι χώρες και όλες οι στρατηγικές θα συμπεριλάβουν την δέουσα προσοχή για τα εργασιακά θέματα και τις σχετικές συνθήκες Πώς σκέφτεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προχωρήσει το θέμα αυτό σε όλες τις στρατηγικές, να συμπεριληφθεί μια σαφή ε, αναφορά για το πώς είναι η κατάσταση στην κάθε χώρα. Κατά δεύτερον, πώς θα εποπτεύουμε την κατάσταση αυτή ανά χώρα. Και προφανώς οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά θέματα. Οι πιο πολλές χώρες έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα εξετάσουμε και τον τομέα της μπανάνας. Θα συμπεριληφθεί δηλαδή σε όλες τις στρατηγικές οι πληροφορίες για το πώς θα γίνει η αξιολόγηση των περιστατικών. Ελπίζω έτσι να απαντώ την ερώτησή σας. Τώρα σε ό,τι αφορά τα πιο γενικά θέματα εμπορίου θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να καλωσορίσω τις θετικές ε, απόψεις της Επιτροπής σας για την Συμφωνία για την πόρο της Μπανάνας. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ιστορική σημασία οι συμφωνίες αυτές. Όχι μόνο επειδή επιλύουν την πιο μεγάλη σε χρόνο διαμάχη στα πλαίσια του ΠΟΕ και να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει σε κάθε στάδιο της ε, διαμάχης αυτής, αλλά η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει ιδιαίτερα το γενικότερο πολυμερές πλαίσιο εμπορίου και ιδιαίτερα και το γύρο της Δόχας. Κατά τρίτον, θεωρώ ότι οι συμφωνίες αυτές ε, ε, θα επιφέρουν μια σταθερότητα, μια προβλεψιμότητα στην αγορά της μπανάνας και γι' αυτό θα βελτιώσουν το γενικότερο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό κλίμα και για τις ε, χώρες ΑΚΕ αλλά και για τους παραγωγούς μπανάνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, οι συμφωνίες αυτής, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικές συμφωνίες, ξέρετε, οι συμφωνίες λοιπόν αυτές προσφέρουν και μία ασφάλεια, μία εγγύηση ότι η προνομιακή πρόσβαση των χωρών ΑΚΕ στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα διαβρωθεί περαιτέρω γιατί στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής συμφωνήθηκε μεταξύ ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής ποια θα είναι τα προϊόντα που θα συμπεριληφθούν στη λίστα διάβρωσης, όπως ονομάστηκε. Θα υπάρξει λοιπόν προνομιακή πρόσβαση σε ό,τι αφορά την μπανάνα και στον μελλοντικό γύρο της Δόχας για να απαντήσω στο ερώτημα για την ενίσχυση του εμπορίου της μπανάνας στις αποκεντρωμένες περιοχές. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε τον κοινωνικό αντίκτυπο και πώς έχει κατάσταση σε αυτές τις αποκεντρωμένες περιοχές. Ωστόσο θεωρούμε ότι τα προβλήματα στην παραγωγή μπανάνας δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων, διεθνών εμπορικών συμβάσεων, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών, εσωτερικών συμφωνιών. Και επίσης να τονίσω ότι κατά τη μεταρρύθμιση της ε, οργάνωσης ε, της κοινή αγοράς για την μπανάνα που έγινε το 2006, τα κονδύλια για τους παραγωγούς μπανάνας στις αποκεντρωμένες περιοχές έχουν αυξηθεί σημαντικά. 278 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το 2007 και μετά. Έγινε επίσης μια μελέτη αντικτύπου και ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάστηκαν ήταν συγκρίσιμο προς τα σενάρια τα δασμολογικά που περιλαμβάνουν τελικά στην συμφωνία για τις ε, μπανάνες. Και τι προέκυψε από την ε, μελέτη αντικτύπου ότι ο αντίκτυπος της απελευθέρωσης του εμπορίου θα πρέπει να έχει ε, περιορισμένο αντίκτυπο. Ωστόσο, κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ της Μανάνας το 2006, ο φάκελος ενίσχυσης των παραγωγών μπανάνας αυξήθηκε. Θεωρούμε ότι έτσι καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες και ο αντίκτυπος των συμφωνιών για την μπανάνα της Γενέβης. Ωστόσο, και θα ήθελα να κλείσω εδώ, να τονίσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά και ασφαλώς και θα λάβουμε δράση αν κρυθεί απαραίτητο. Και τέλος τέλος, να υπογραμμίσω κάτι άλλο, να μην το πω σφάλμα, πρόκειται για μια πτυχή που δεν θεωρούμε ότι είναι απολύτως ορθή σε ό,τι αφορά την αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Καταρχάς, ε, οι ζώνες ε, καλλιέργειες του 114 μιλάμε για το 2017 θα είναι η πιο πρώιμη ε, ημερομηνία. Γιατί αν υπάρξει δύο χρόνια καθυστέρηση, αυτό θα αφορά και την αγορά της μπανάνας. Κατά δεύτερον, στα πλαίσια της Συμφωνίας της Γενέβης, την οποία και πραγματευόμαστε σήμερα, το όριο του 75 ευρώ ανατόνο είναι λίγο παραπλανητικό, γιατί αυτό αναφέρεται στι διμερείς συμφωνίε, τι οποίε θα πρέπει να εξετάσουμε υπό διαφορετικό πρίσμα και σε διαφορετικό πλαίσιο. Ο κ. Γκούρεντ, λέει, πρόεδρο, έχει το λόγο και να ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτέ τι επιπλέον ε, εξηγήσει και εγώ τώρα θα ήθελα να δούμε τα πράγματα ω εξή Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ολοκληρώσουμε τα του ψηφίσματος πριν τη συνάντηση κορυφής. Τι θα μπορούσαμε σε ένα τέτοιο ψήφισμα να εντάξουμε. Έχουμε την προβληματική τη γνωστή, γιατί μας λέει η Κομισιόν ότι όσον αφορά τις εμπορικές προτιμήσεις είμαστε απομονωμένοι. Και εσείς είπατε όσον αφορά κάποιες ε, ευρωπαϊκές χώρες ότι υποφέρουν σε σχέση με αυτή την ε, ε, ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχει αυτό το βεθύλιο. Οπότε θα μπορούσαμε να συμμαχίσουμε με τις αφρικανικές χώρες. Μιλούμε για 80 χώρες. Και βλέπετε ότι γίνεται. Έχουμε τις αναδυόμενες χώρες και το G90 και οι Αφρικανοί εξαπατώνται. Τους κορυδεύουν επίσης θα πρέπει να σας πω αυτό το οποίο ήταν η αρχή του προβλήματος. Η Βραζιλία και άλλες χώρες θέλουν να πάρουν το καλύτερο κομμάτι της αγοράς. Και έτσι κάποιες αυξημένες χώρες ρίχνουν κάποιες άλλες. Εμείς όμως θέλουμε να τονίσουμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι πολιτικό το, επίπεδο στο οποίο θέλω να το αναδείξουμε αυτό το ζήτημα και μας δίνει το ευκαιρία τώρα να το κάνουμε. Και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαι σύμμαχος μας σε αυτή την ε, προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω θα πρέπει να συγκρίνουμε τις προσπάθειές μας μέχρι ότου πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Να, μια αξία που μπορούμε να, να δώσουμε στα πλαίσια Εξωτερικής Πολιτικής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Προθεσμία για την ε, κατάθεση είναι 27 Οκτωβρίου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 9 ε, Νοεμβρίου τις τροπολογίε. Τώρα, η ενεργειακή πολιτική της Παγκοσμίας θα συζητήσουμε μια προφορική ερώτηση και ένα σχέδιο ψηφισματο. Όπω ίσω ήδη γνωρίζετε, η Παγκόσμια Τράπεζα τώρα σχεδιάζει την ενεργειακή τη στρατηγική. Θα εγκριθεί το 2011 μετά από μια διαβούλευση με του διάφορου εμπλεκομένου και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προτινόμενη στρατηγική για τον ενεργειακό τομέα πρόκειται να καθορίσει τα μέσα με τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τι αναπτυσσόμενες χώρε. Διπλό είναι ο στόχο. Πρώτα-πρώτα να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα στην ενεργεία, ενέργεια στην αυτάρκεια τη, όσον αφορά την προμήθεια. Και από την άλλη μεριά θα έχουμε καλύτερη πορεία προ ένα μοντέλο το οποίο να είναι βιώσιμο βάση οικολογική και αξιοποιώντα ενέργεια. Βλέπουμε επομένω πόσο σημαντική είναι η ενέργεια για την βελτίωση της, του βιωτικού επίπεδου αυτών των χωρών. Πρέπει να πετύχουμε του στόχου τη χιλιετία, αλλά θα πρέπει αυτή η στρατηγική να είναι στοχευμένη και να γίνεται με συντονισμό με τις άλλες χώρες. Έχουμε αυτή την προφορική ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος με τα οποία η Επιτροπή μας θέλει να τονίσει εξή. Πρώτα-πρώτα ότι χρειάζεται να υπάρχει ανεφοδιασμός των ε, κοινοτήτων, των χωριών στην ε, Ήπεθρο και αυτό να αφορά τις ε, ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και στη συνέχεια θα πρέπει να στηρίξουμε τη στρατηγική της τράπεζας όσον αφορά τις επενδύσεις που σιγά σιγά θα μειώσουν τη χρήση του άνθρακα και του διοξιδίου του, του άνθρακα. Και σε σχέση με αυτό έχουμε συντάξει την προφορική ερώτηση αλλά και το σχέδιο του κειμένου. Έχετε τώρα εσείς συναδελφοί το λόγο. Ποιος θέλει το λόγο. Νομίζω ότι υπάρχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κύριο Σάντερ Σίπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε για το ότι μα δίνει το δικαίωμα να σα μιλήσουμε σήμερα. ως Παγκόσμια Τράπεζα. Είμαστε σε επαφέ και με την Επιτροπή σα και με άλλε επιτροπέ και φέρουμε πάντα την πολιτική μα στις Βρυξέλλε και στο Κοινοβούλιο. Εσείς και ο Γιώ Λάινεν είναι συμπρόεδροι. Είναι τιμή αυτό για μας και το συζητήσαμε ήδη το 2009. Φέρουμε τη στρατηγική μας εδώ τον Μάιο του 2010. Η ενεργειακή πολιτική συζητήθηκε στις 27 Μαΐου με πολλούς ενδιαφερόμενους, συμπεριβαίνουμε και μεταξύ και μερικών ευρωβουλευτών. είχαμε το σχέδιο ψηφίσματος. Θεωρούμε το σχέδιο ψηφίσματος πολύ ενθαρρυντικό. Και επισημαίνω ότι η στρατηγική μας είναι ένα δυναμικό, μια δυναμική διεργασία. Έχουμε τελειώσει την πρώτη φάση, όπως τη λέμε upstream, με τις κύριες ιδέες και το πλαίσιο της στρατηγικής μας και τώρα περνάμε στην φάση 2. Γράφουμε τη στρατηγική και θα περάσουμε σε μια νέα φάση διαβουλεύσεων. Αναφέρω από το σχέδιο ψηφίσματό σας όπου καλείται να ενθαρρυνθεί η Παγκόσμια Τράπεζα η στρατηγική της να έχει προγράμματα με χαμηλό ίχνος άνθρακα και καινοτόμα χρηματοδότηση και θεσμική ανάπτυξη. Προσθέτω ότι δεν χάνουμε χρόνο, κινούμαστε ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή με πολλαπλές επενδύσεις και έχουμε μια ομάδα για την περιοχή Μέση Ανατολή Βόρεια Αφρική θα θεί εδώ να διαπραγματευτεί με την Κομισιόν και άλλους εταίρους ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για ανανεώσιμες πηγέ ενέργειας και πιο συγκεκριμένα ηλιακή ενέργεια στη Βόρεια Αφρική. 6 δις δολάρια είναι η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την ευκαιρία που μας δώσετε να σας μιλήσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Κομισιόν τώρα. Ο κύριος Λουί Κώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο συνάδελφος από την Παγκόσμια Τάπαζα, Αυτή τη στιγμή συντάσσεται η στρατηγική μετά από την πρώτη φάση διαβουλεύσεων, το πρώτο εξάμεινο. Είχαμε συνάντηση όλων των υπηρεσιών στις 27 Μαΐου. Κάναμε σχόλιο ως Κομισιόν. Έχουμε μία σύνοψη, ξεκινώντας την φάση υπαριθμών 2 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μερικές από τις υποδείξεις μας υπάρχει σε αυτή την σύνοψη. Θετικό αυτό. Ελπίζουμε να μείνουν και στο τελικό κείμενο. Γιατί έτσι το κείμενο, το έγγραφο βελτιώνεται. Στην Ένωση έχουμε μια ενεργειακή πρωτοβουλία για την εξάλληψη της φτώχειας και την ε, βιώσιμη ενέργεια μετά το Johannesburg του 2002 ξεκίνησαν αυτά, αυτή η πρωτοβουλία με τακτικές συναντήσεις κρατομελών, κομισιών και ελπίζουμε να το έχουμε στην σε διάταξη την επόμενη φορά, αυτή τη στρατηγική δηλαδή, το τελικό κείμενο εννοώ της Παγκόσμιας Τράπεζας για συντονισμό. ετέθη ερώτημα επιλογές ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Θα τις προωθήσουμε ή όχι. Το 2007 στη Λισαβόνα ξεκίνησε η εταιρική σχέση Ένωση Αφρική. Μπορεί να μας πείτε ότι επικεντρώμε την προσοχή μας στην Αφρική και ξεχνάμε άλλα τμήματα της Ιφιλίου. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά με την εταιρική αυτή σχέση Πρόσφατα οργανώσαμε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου με 26 υπουργούς ενέργειας και επιτρόπους από Ευρώπη και Αφρική και εκεί εγκρίθηκε στόχος για την Αφρική διότι 2020 για τις ανανεώσιμες ενέργειες και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επίσης ξεκίνησε στόχος 2020 η πρώτη φάση 2010-2013. Η Κομισιόν θα είναι ο πρώτος που θα συμβάλλει στη φάση αυτή για το πρόγραμμα συνεργασίας για τις ανανεώσιμες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας θυμίζω ότι και το ερώτημα και η πρόταση ψηφίσματος θα εγκριθούν το Δεκέμβριο στην Επιτροπή μας και μετά θα τεθούν προς ψηφοφορία στην Ολομέγεια του Ιανουαρίου. Προθεσμία για τροπολογίες 15 Νοεμβρίου. Και το τελευταίο σημείο για σήμερα είναι η γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Γεωργίας για τη Γεωργία και το Διεθνές Εμπόριο. Η κυρία Τόγια, η συγγήτρια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Η έκθεση αφορά μια έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Γεωργίας και ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή ΙΝΤΑ για το Διεθνές Εμπόριο και Γεωργία της Ένωσης. Επειδή έχουμε τις περίφημες 1000-1500 λέξεις, προσπάθησα σε αυτή τη γνωμοδότηση να μείνω στα βασικά θέματα ή το βασικό θέμα και με τις τροπολογίες που εγώ θα προτείνω και οι συνάδελφοι, θα συμπληρώσουμε και θα εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο της γνωματότησής μας. Το έγγραφο ξεκινάει από μια ανάλυση της κατάστασης που όλοι την ξέρουμε. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία κάνει την Ευρώπη μια από τις πιο μεγάλους εισαγωγείς γεωργικών προϊόντων και η Ένωση έχουμε σημαντική μείωση της εξαγωγικής μας ικανότητας. Παρά τα συστήματα επιδοτήσεων και ενισχύσεων στις εξαγωγές, το οποίο υφίσταται επί σύστημα, αλλά το σύστημα αυτό από μια μεριά δεν βόηθησε τις εξαγωγές μας, γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη μείωση, και απ' την άλλη δημιούργησε dumping και στρεβλώσεις σε σχέση με άλλες χώρες που βρέθηκαν σε τελείως άνισες συνθήκες λόγω των ενισχύσεων των εξαγωγών μας. Και άλλη επιπλέον στρέβλωση, τότε συχνά δημιουργούμε δύσκολε καταστάσεις για τις λιγότερα αναπτυγμένε χώρες που δεν μπορούν να βγάλουν τα προϊόντα του στην αγορά. Μερικές φορές βοηθήσαμε χώρες όπου με τα χρόνια αυξάθηκε η οικονομία του και να παράγουν και να εξάγουν στη διεθνή αγορά. Βραζιλία, Κίνα, χώρες με ψηλό δυναμικό που ενισχύονται επιπλέον από τα εσφαλμένα μέτρα μας. Είναι ευκαιρία να επικαιροποιήσουμε τη θέση μας. Με την αναθεώρηση της ΚΑΠ που συζητιέται και το οποίο την άνοιξη του Κοινοβούλου είχε πάρει θέση και δεύτερο σε σχέση με το ότι σταμάτησαν οι διαπραγματεύσει στις πολυμερείς σχέσεις και έχουμε ανταυτού διμερείς συζητήσεις και συμφωνίες στο παγκόσμιο εμπόριο και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που αφορά τη γεωργία και το παγκόσμιο εμπόριο. Το βασικό σημείο είναι αυτό. στο κείμενο της Γεωργίας δίγεται καν υπενιγμός στον προβληματισμό για τη σχέση Γεωργία με τη διεθνή συνεργασία και το ρόλο της Ένωσης για την ανάπτυξη στον κόσμο. Ούτε καν υπενιγμός, ενώ το έγγραφο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου που μιλάει για την εξωτερική δράση της Ένωσης εμπορικά αναφέρεται στο ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης αφορά πολιτικές ε, ανάπτυξης και βοήθεια για την ανάπτυξη. Είναι και αυτό εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Το κύριο θέμα λοιπόν είναι ότι δεν αρκεί να μιλάμε για τη συνοχή που πρέπει να υπάρχει μεταξύ γεωργία και διεθνές εμπόριο. Χρειάζεται μια διεθνής ακολουθία στις πράξεις μας Και αυτό πρέπει να μπει στη γνωμοδότηση. Γιατί η δραστηριότητα της Ένωσης εσωτερικά και εξωτερικά πρέπει να διέπεται από μία ανακολουθία. Και όλα αυτά δεν είναι περιτά, πρέπει να τα επισημάνουμε. Δεν είναι δευτερεύοντα. Πρέπει επίσης να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει λογική ακολουθία και απορρέει αυτό και από τις συνθήκες και από τις πράξεις μας και είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη της γεωργίας και των τροφίμων Όλοι το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, η οικονομική κρίση έπληξε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και την παραγωγική τους ικανότητα, η κρίση λόγω της αλλαγής του κλίματος πλήττει τις χώρες αυτές και όλα, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στον αναπτυγμένο κόσμο λόγω της αλληλεξάρτησης. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτή η λογική ακολουθία. Θέλω μια γεωργική πολιτική που να είναι βιώσιμη και δίκαιη. Με ανταγωνιστικό εμπόριο, μεν, αλλά ικανή να δημιουργεί πιο δίκαιες σχέσεις όσον αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων γενικότερα. Ε, πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο κύριε Γκέρεντς. Ναι, γιατί θέλω να πω κάτι για την εκθέση Τόια. Ορθά μας είπε ποιες είναι οι επιπτώσεις από τις εξαγωγικές επιδοτήσεις όσον αφορά τη γεωργία και τις εμπλησόμενες χώρες. Θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει περισσότερο από το το 2000 φτάναμε στα 10 δις ευρώ. Το 2008 κατεβήκαμε στα 400 και κάτω. Επομένω είναι πάρα πολύ θετικό αυτό και δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Και διαδεσμευτήκαμε στην Τόχα να καταργήσουμε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις και πιστώσεις για τις νέες εμπορικές συμφωνίες. Αν δεν κάνω λάθος δεύτερο σημείο που θέλω να σας αναφέρω. Όσον αφορά το ρόλο μας για τις εμψωμένες χώρες θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι έχουμε το dumping της Κίνα σε σχέση με αυτά τα οποία κάνει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως έχουμε φτάσει όντως κατά υποτίμηση του κινέζικου νομίσματος. Ενώ εμείς κάνουμε τον ενάρετο και πρόκειται για έναν νομισματικό ε, πόλεμο και τώρα διακυμαίνεται ελεύθερα στην παγκοσμία αγορά το One, το κινέζικο νόμισμα και δεν είναι μόνο η Κίνα που κάνει τέτοια πολιτική, θα πρέπει να δούμε τι κάνουν και οι άλλοι. Ε, και τέλος πάντων σε σχέση με αυτό το που έχουμε κάνει εμείς στο παρελθόν να το εξετάσουμε. Τώρα για αυτά τα οποία προτείνεται να ενθαρρύνουμε δηλαδή μια θεαματική μείωση των δασμών που αφορά τις εισαγωγές προϊόντων των εμψωμένων χωρών του Νότου. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση και αντίφαση με αυτό το οποίο πρότεινα εγώ στη δική μου έκθεση που συζητήσαμε προηγουμένω. Που θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, προτιμησιακή εμπορική πολιτική με τι χώρε αυτές. Ενώ εσεί προτείνετε αυτή την διαφοροποίηση. Θα πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς είναι δυνατόν αυτή η πρόταση να ενταχθεί στην θέση μας. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Επιτροπή μας συζητάει και καταρτίζει την γνωμοδότηση αυτή για τα θέματα αυτά, γιατί φυσικά η γεωργία είναι ένας από τους κατεξοχήν τομείς όπου υπάρχει ασυνέπεια και πρέπει να επεμβούμε και φυσικά είναι σημαντικό το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξουν τέτοιες ε, ε, επιδοτήσεις. Ε, συζητήθηκαν πολλές φορές στο παρελθόν και φυσικά το τι γίνεται στην Ευρώπη επηρεάζει και τις παγκόσμιες τιμές γιατί παράγουμε μάλλον ε, διαθέτουμε φτηνά προϊόντα επειδή επιδετούνται στις αγορές. Για παράδειγμα, τα γαλακτοκαμικά, οι ντομάτες, το κατεψυγμένο κοτόπουλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να παρακολουθεί την κατάσταση και να παρεμβαίνει στη συζήτηση αυτή. Και αυτό δεν ε, συμπεριλαμβάνει μόνο την Επιτροπή Γεωργίας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την εξωτερική πτυχή της μεταρρυθμίσης της ΚΑΠ. Μία ιδέα θα ήταν λοιπόν να γίνει μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Γεωργικής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι προγραμματίζεται αυτό. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, συμφωνώ με τα περισσότερα στοιχεία τα οποία ανέφερε η κυρία Τόγια και χαίρομαι ιδιαίτερα που το θέμα του PCD e αναφέρεται στην έκθεση αυτής. Το πρόβλημα, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι μόνο οι άμεσες επιδοτήσεις εξαγωγών, αλλά και οι έμεσες επιδοτήσεις. Η έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΑ αναφέρει ότι παράγει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αναφέρονται στις εισαγωγές που κάνουμε. Και πώς επηρεάζουν, για παράδειγμα, το, την αλλαγή του κλίματος, την ε, βιοπικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει κυρίως μεταποιημένα προϊόντα και αυτό φυσικά έχει και ένα κάποιον αντίκτυπο και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Τι γίνεται, για παράδειγμα, το 2015 θα ε, ε, έχουν ε, καταργηθεί οι ποσοστώσεις για τα χαρακτηροκομικά, για τα γάλα. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλές περιπτώσεις κάνει υπερβολικές υποχωρήσεις σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσει. Δεν ξέρω αν σύμφωνο. Θεωρώ, και αυτό καταδεικνύεται και από τους γύρους της Ντόχα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει παίξει ακόμα το ρόλο που θα έπρεπε. Κάτι άλλο που θα μας απασχολήσει για το μέλλον της ΚΑΠ. Τα τρόφιμα τα οποία ε, εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οι χώρες που τα εξάγουν να είναι σε θέση πρώτα να θρέψουν τον ίδιο τους τον πληθυσμό. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. La parole est maintenant à la Commission. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Συμβένας από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα την ε, εισηγήτρια. Δεν έχω και πολλά να σας πω. Γιατί ο κύριος Γκέρενς είπε τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να σας πω εγώ. Όσον αφορά πρώτα πρώτα τις εξαγωγές επιδοτήσεις. Όντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί στα πλαίσια του γύρου της Ντόχα να καταργήσει πάσα ενίσχυση εξαγωγική. Και παράλληλα να καταργήσει παντός άλλου είδους επιδότηση. Και αυτό όσον αφορά και τι αναπτυσσόμενε χώρε, όσον αφορά δηλαδή την διατροφική ενίσχυση, όσον αφορά τι ε, κρατικέ επιχειρήσει, το κρατικό εμπόριο δηλαδή που αφορά τι χώρε αυτέ. Εμεί θα τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση. Και θέλουμε το 2013 να υλοποιηθεί αυτό το οποίο είπαμε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο αφορά τις επιστροφές τις εξαγωγικές, είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες εξαγωγικές επιστροφές, περισσότερες από αυτές έχουν καταργηθεί και πέρσι για κάποια περίοδο προσωρινά ίσχυσαν κάποιες τέτοιες εξαγωγικές επιστροφές όσον αφορά τα γαλακτοκομικά. Σα υπενθυμίζω ότι είχε πέσει εντυπωσιακά η πτώση των γραπτοκομικών κατά 60% όμως πάρα αυτά δεν θελήσαμε να συμπληρώσουμε τη διαφορά μεταξύ της ε, τιμής αυτής και της παγκόσμιας τιμής απλώς εν μέρη να το κάνουμε αυτό και μόλι η ευρωπαϊκή ε, αγορά βρήκε την ισορροπία της καταργήσαμε και αυτό το μέτρο. Τρίτον, Βεβαίως και υπάρχει θέμα υποκατάστασης και αντικατάστασης και όταν δεν είμαστε εμείς παρόντες η τοπική παραγωγή μας αντικαθιστούν για μας ή υποκαθιστούν για παράδειγμα στην Ιγυρία. Για την Ιγυρία και το Γάλα η Νέα Ζηλανδία μας αντικατέστησε. Τελευταίο τώρα σημείο, σαν το σημείο υπερθμόνου. 5 για την κατάργηση των δασμών για τις αντισόμενες χώρες. Για όλες τις χώρες ε, ΑΚΕ έχουμε ανοίξει τελείως τα σύνορα. Άρα μπορούν να εξαγάγουν χωρίς ποσοτικό περιορισμό, χωρίς να υφίστανται δασμούς όσον αφορά την αγορά μας. Και αυτός και για όλα τα γεωργικά προϊόντα χωρίς εξαίρεση. Οι χώρες ΑΚΕ άλλωστε είναι από τι πτωχότερες στον κόσμο. Βλέπετε επομένω που έχουμε ανοιχτή πολιτική όσον αφορά αυτές τις ε, φτωχές χώρες. Εν κατακλείδη, σας αναφέρω ότι ξεκίνησαμε μια ευρεία διαβούλευση για την ΚΑΠ. Για μετά το 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία θα κάνουμε μια μελέτη επιπτώσεων, θα κάνουμε μια ανακοίνωση για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να επανεξεταστούν. Και θα κατεβάσουμε τις προτάσεις μας του χρόνου. Merci beaucoup, Monsieur Olthoff de DG Développement. Non, vous ne demandez pas la parole. D'accord. Ούτε ο κ. Olthoff θέλει το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη. Για το όμως θέλει να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν και την συμβολή των συναδέλφων θα περιμένω. Όσον αφορά τη μείωση των επιδοτήσεων, είπα ότι μας αρέσει η μείωση αυτή και τα δύο νούμερα που ανάφερε στην Κέρνς το αποδεικνύουν το πόσο σημαντική ήταν αυτή η μείωση. Ζητάμε να συνεχιστεί αυτή η κίνηση. Αυτό είναι το κείμενό μου, είναι ένα πρώτο κείμενο. Φυσικά θα γίνουν διορθώσεις και θα μπουν και νέες ιδέες. Και στο σημείο 5 πρέπει να είμαστε συνεπείς. Από τη μία μέρα μειώθηκαν οι δασμοί και από την άλλη μεριά να κάνουμε αυτό που είπαμε. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται α συνεργαστούμε και με τροπολογίες και με προσωπική του συμβολή, θέσεις. Αυτό και είμαι υπέρ αυτού και με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Πρόεδρος, προθεσμία για τροπολογίες 9 Νοεμβρίου, 12 η ώρα. Ψηφορία στην Επιτροπή μας στις 9 Δεκεμβρίου. διάφορα. Τίποτα. Η επόμενη συνεδρίασή μας στις Βρυξέλλες 8 Νοεμβρίου στις 3 η ώρα και την 3η 9 Νοεμβρίου 9 Πέρασε. περας